La seduta è ripresa. Procediamo ora. Η σύνοδος συνεχίζεται. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Πρώτη, η έκθεση του κυρίου Παντζέρη για την Συμφωνία Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλγερίας για τις γενικές αρχές της συμμετοχής της Αλγερίας στα προγράμματα της Ένωσης. Η ψηφοφορία είναι ονομαστική. Η ψηφοφορία άρχεται. πέρα τη πληροφορία. Εγκρίνεται. Η έκθεση συγχαρητήρια στον κύριο Παντζέρη. Έκθεση Τομά. Βορειοανατολικό Ατλαντικό από θέματα βαθέων υδάτων και αλλιέ σε διεθνή υδάτα. Τροπολογία 1 για θέση Συμβουλίο 1. Άρχεται η ψηφοφορία με, και είναι ονομαστική. Πέρας. Η τροπολογία απορρίφθηκε, οπότε η πράξη εγκρίνεται βάσει της, της που έχει ε, συμφωνηθεί μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Περνάμε τώρα στην έκθεση Corbett. Διαδικαστικό από τον κύριο Φερέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το γεγονός ότι έχουμε μπροστά μας μια έκθεση που αυτή τη στιγμή ε, έχει πάνω από 400 τροπολογίες σημαίνει ότι πόρο απέχουμε από το να έχουμε οποιαδήποτε συνένεση. Η διαδικασία αυτή δεν έχει